Ευχαριστούμε την Επίτροπο Ρέντινγκ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση λοιπόν. Έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος και θα ακολουθήσει άμεσα η ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω. Έχουμε ένα διαδικαστικό θέμα από ποιον. Ένα αίτημα, Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και για τα τρία ψηφίσματα. Ευχαριστώ. Herr Έληξε η προθεσμία σήμερα το πρωί, συνάδελφε. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι έχουμε λάβει μια πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την εσωτερική αγορά, την ηλεκτρονική επικοινωνία και για τροποποίηση της οδηγίας 2002-2001 και 2021 και του κανονισμού 1211. Αυτά είναι έγγραφα τα οποία δίδονται στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας, Επιτροπή Πολιτισμού, Νομική Επιτροπή, Επιτροπή Δικαιοσύνης, Εσωτερικής Αγοράς Προστασίας των Καταναλωτών, Περιφερειακή Πολιτική. Θα είναι οι συνεργαζόμενες επιτροπές. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Καταρχήν για έξι ψηφίσματα όσον αφορά την κατάσταση στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένα κοινό ψήφισμα, παράγραφος 6 του αρχικού κειμένου, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου, υπέρ, κατά, αποχές, ομόφωνα εγκρίνεται. Τώρα, ψηφοφορία για πέντε προτάσεις ψηφίσματος για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έχουμε το κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων. ψήφισμα για το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα, καθώς βλέπω. Και τέλος ψήφισμα για την κατάσταση στο Μπαχρέιν. Εδώ έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος και ένα κοινό ψήφισμα τεσσάρων πολιτικών ομάδων με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για το του ψηφίσματο. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Με 7 αποχές ομόφωνα εγκρίνεται. Τα πρακτικά θα είναι έτοιμα στην έναρξη της επόμενης συνόδου του Κοινοβουλίου και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και θα στείλουμε σε αυτούς τους οποίους απευθύνονται τα ψηφίσματα αυτά. Σας εύχομαι